Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Βλέπω ότι παρά τις ελαφρές ε, χιονοπτώσεις, πολύ τα καταφέραμε να έρθουμε στο Κοινοβούλιο. Το σπίτι μου μπροστά είχε 40 εκατοστά. Εδώ ίσως είναι λίγο λιγότερο το χιόνι. Κάθε περιοχή είναι διαφορετικά το χειμώνα και διαφορετική προετοιμασία κάθε φορά σε κάθε περιοχή. Πάντως ε, ωραία είναι οι Βρυξέλλες με το χιόνι, ε, μας αλλάζει την καθημερινότητα. Είμαστε αρκετοί συνάδελφοι, μπορούμε να ψηφίσουμε. Είχαμε προτείνει να ξεκινήσουμε με, την, ε, με το σημείο 12 της μέσης ε, διάταξης, ε, με την έκθεση Μπερλάτο για ένα τέταρτο. Μετά θα έρθει ο πρόεδρος Μπούζεκ για μια σύντομη συνάντηση και είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε στα 20-25 λεπτά περίπου να ακούσουμε τον Πρόεδρο και μετά κάθε πολιτική ομάδα εν συντομία ένα-δύο λεπτά να λάβει το λόγο και μετά να ακολουθήσει η ψηφοφορία για το σημείο 11, για το σημείο της κυρίας Μαρίζα Ματίας για την όσο του Αλτσχάιμερ που έχουμε και τροπολογίε. Ελπίζω θα τα καταφέρουμε λοιπόν με αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν την έκθεση του Σέργιο Μπερλάτο αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επιστηστικής ασφάλειας. Να ψηφίσουμε για την πρώτη τροπολογία. Αρσένης Λεπάς Πυρίλιο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να βάλω και... Τροπολογία 3. Φερέιρα. Τζομαρία Ουτζιά. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Τζομαρία ουτζιά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Φερέιρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Φερέιρα Τζομαρία Ούτζιας. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Τζομαρία Ούτζιας Τζοάου Φερέιρα. Ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 πυρίλιο κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 Ελένα Αντωνέσκου ψήφι υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 9. Άλλη μια φορά αρχίζει η ψηφοφορία, επαναλαμβάνουμε. Άλλη μια φορά. Ζητώ συγγνώμη. Πέρασε Η ψηφοφορία. 22 υπέρ, 25 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 11. Τζομαρία Ούτζε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10, Ροβάνα Πλάμ, ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12, Φερέιρα Αρσένης, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Έστειο Ντελάνγκε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει το τρίτο τμήμα. Έχουμε και ένα τέταρτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Πάλι κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Να το ελέγξουμε. 20, πρώτο τμήμα, ελέγχουμε. Έλεγχος για το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 20. Να και η κάρτα του κ. Γιώργενσεν. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ναι, ναι, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. Τροπολογία 23. Γκαρντίνη. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27 James Nicholson. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται, αλλά μάλλον να το ελέγξουμε. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 28 Λεπάζιο Μαρία Ουτζιάς. Εδώ έχουμε... Μια προφορική τροπολογία στην τελευταία πρόταση δεν θα λέει and development Δεν θα λέει development στο τέλος, θα λέει μόνο agricultural practices. Μόνο αυτό. Με την προφορική τροπολογία λοιπόν ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ της 28. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν βοήθησε ούτε η προφορική τροπολογία. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές.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 Πέρας της ψηφοφορίας. Υπέρ, σαφώς. Εγκρίνεται λοιπόν. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 ψηφοφορία κατά τμήματα. Στο πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, Οι πράσινοι δεν ψηφίζουν. Ψηφίζετε. Ναι, όχι, τι ψηφίσατε. Να ελέγξουμε λοιπόν τη 44. Πρωί-πρωί τα μπελιάζεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Ναι, κατανοώ ότι παρότι καθυστερήσατε, κάνατε, παίξατε σημαντικό ρόλο και κάνατε τη διαφορά στην ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Μετά περνάμε στην 45 πυρίλιο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 αποσύρεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές με την ίδια πλειοψηφία και πάλι εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 Ροβάνα Πλάμ κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε για την 54. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται επίσης. Περνάμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. 44 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, 6 αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Μπερλάτο. Ο πρόεδρος θα έρθει όπου να είναι. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Μαρίζα Ματίας να μας πει τρία-τέσσερα λεπτά δύο λόγια για τις συμβιβαστικές τροπολογίες. για να δούμε πώς έχει η τωρινή κατάσταση των πραγμάτων. Μπορεί η κυρία Μαρίζα Ματίας να μας παρουσιάσει την κατάσταση για την έκθεσή της και μετά θα έχουμε την ε, συναντήση με τον πρόεδρο Μπούζεκ. Κυρία Ματίας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Απλώς να κάνω μια σύντομη παρουσίαση ε, και εισαγωγή για να δούμε τι θα ψηφίσουμε και ποιες είναι οι συμβαστικές τροπολογίες στις οποίες καταλήξαμε. Τα όρια τα οποία είχαμε ορίσει για την έκθεση αυτή σήμαινε ότι ένα μεγάλο τμήμα του περιεχομένου αυτής της έκθεσης έπρεπε να προέρθει από τις τροπολογίες. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους, όλους τους συναδέλφους, όχι μόνο τους σκιώδεις εισηγητές, αλλά και όλους τους συναδέλφους, διότι ακριβώς με τις προτάσεις τους εμπλούτησαν την έκθεση και στο τέλος... Και στο τέλος καταλήξαμε σε μια μεγάλη σειρά τροπολογιών 103 ενοποιημένες τροπολογίες έχουμε και 16 περίπου συμβιβαστικέ. Μέσω αυτών των ε, συμβιβαστικών τροπολογιών, αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα βασικά θέματα, στα κέρια σημεία της έκθεσης και η θέλαμε να τονίσουμε την ε, ε, σημασία ε, που έχει η πρόορη διάγνωση, η πρόληψη επίσης. Αυτό είναι ένας από τους στόχους μας. Επίσης θέλησαμε να τονίσουμε τη σημασία της συνεργασίας που έχει, ε, τη σημασία που έχει συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει να έχουμε μια συνολική, μια σφαιρική, ε, ένα σφαιρικό συντονισμό των δραστηριοτήτων και να μην έχουμε κατακαιρματισμένες ενέργειες πρέπει να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα, να διδαχτούμε από τα παθήματα του παρελθόντος, γιατί ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η νόσος αυτή πλήττει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, του ευρωπαϊκού πληθυσμού και θα πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις πρακτικές, να εφαρμόσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόσουμε σε όλη την Ευρώπη. Ένα άλλο σημαντικό θέμα επίσης είναι η έρευνα και ε, προσπαθήσαμε να επωφεληθούμε από τις πρόσφατες ε, εξελίξεις γιατί υπάρχουν και κάποια κενά στις επιστημονικά δεδομένα ε, σε αυτόν τον τομέα. Όσον αφορά παραδείγματο χάρη τα αίτια, τα συμπτώματα, ε, κάποιες, άλλες, κάποιες πτυχές της άνοιας μας είναι τελείως άγνωστες. Απ' την άλλη πλευρά έχει γίνει πάρα πολλή έρευνα βέβαια. Γι' αυτό θα πρέπει να εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας στον τομέα της έρευνας σε όλα τα κράτη. Και το έχω τονίσει κι εγώ ότι πέραν της φαρμακολογικής έρευνας πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλους τομείς. Και αυτό εκφράζεται στις ε, ε, συμβαστικές τροπολογίες. Επίσης το υπάρχει και το θέμα της αξιοπρέπειας του ασθενούς αλλά και, την, ε, και υποστήριξη των συγγενών και των οικείων του, του ασθενούς. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι και ο ασθενής ο ίδιος. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Απλώς να, τον, να πούμε ότι ε, θελήσαμε να τονίσουμε κάποια σημεία περισσότερο. Γι' αυτό ευχαριστώ και τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες. Ε, προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη μας όλες τις προτάσεις που ακούστηκαν. Πιστεύω ότι η συνεισφορά όλων ήταν ιδιαίτερα θετική και όλες οι συνεισφορές εμπλούτησαν και βελτίωσαν την αρχική έκθεση και ελπίζω ότι οι συμβαστικές αυτές τροπολογίες αποδίδουν πιστά το πνεύμα των ε, συναδέλφων όταν έκαναν τις προτάσεις τους. Και τους ευχαριστώ όλους για μια εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τη Μαρίζα Ματίας για τις παρατηρήσεις που μας έκανε για τις συμβαστικές τροπολογίες. Έχετε άλλες ε, παρατηρήσεις ή σχόλια από αυτού οι αντιρρήσεις. Δεν βλέπω να υπάρχει αντίδραση. Ο πρόεδρος πότε έρχεται, πρέπει από λεπτό σε λεπτό να φτάνει. Στις 9.30 έρχεται ο πρόεδρος. Να περιμένουμε, απλώς ας περιμένουμε. Για να μην αρχίσουμε την ψηφοφορία και τη διακόψουμε. Αλλά και να περιμένουμε πάλι δεν έχει νόημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Τηλεφωνήσαμε για να δούμε πότε έρχεται ο πρόεδρος και έρχεται. Θα διακόψουμε όταν έρθει. Λοιπόν, ξεκινάμε με την ψηφοφορία. Παράγραφος 1, τροπολογία 75 της Μαρίζα Ματίας της ίδιας ψήφι υπέρ. Συμβιβαστικές ψηφοφορίες. Συμβιβαστική λύση 9 για την πρώτη παράγραφο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Μετά στη δεύτερη σελίδα, Κριστίνα Γκουτιέρες Κορτίνας, 78 ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 79 Αντωνέσκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά περνάμε στην συμβαστική τροπολογία 10 για την παράγραφο 2. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά προχωράμε με την 89 του κυρίου Σκυλακάκη. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται επίσης. 90 με μια προφορική τροπολογία στο δεύτερο τμήμα, αλλά έχουμε κατά τμήματα, ψηφίζουμε πρώτα το πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. 91. Νέσα Τσίλντες, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 για την παράγραφο 3, ψήφι υπέρ. Κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. 97. Φρεντερίκ Ρίς. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 για την παράγραφο 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 101. Για να κουδάκι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102. Για να κουδάκι και πάλι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές. Αυτό πρέπει να το ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία, την 108 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13 για την παράγραφο 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την επόμενη ψηφοφορία κατά τμήματα, πρώτο τμήμα για την 115, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Να είμαι στην 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχει έρθει ο πρόεδρος όμως. Κάνουμε μια σύντομη διακοπή για να περάσουμε στη συνάντηση με τον πρόεδρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την τιμή και τη χαρά να καλωσορίσω τον Πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Μπούζακ, που γνωρίζει τα θέματα για την αλλαγή του κλίματος και στην προηγούμενη θητεία ήταν μέλος της Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή και συνόδευσε και την αντιπροσωπεία μας κατά τις εργασίες μας στην Κοπενχάγη πέρυσι. Ο Πρόεδρος μας υποστηρίζει, υποστηρίζει τη δουλειά μας, είναι θετικό αυτό για μας και την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο Είχαμε και ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την, για την διάσκεψη στη Κανκούν. Υπήρχαν πολλές ε, διαφορές, αλλά υπήρχαν και πολλές κοινέ θέσεις ε, εδώ σε εμά, ε, πέρα από κομματικές αντιπαραθέσεις και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο Μπούζεκ για να μας κάνει κάποιες παρατηρήσεις προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος για το θέμα αυτό, για την Κανκούν, για την προστασία του κλίματος και τον συνολικό τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, Καλημέρα, ε, συνάδελφοι. Ζητώ συγγνώμη γιατί διατάραξα την, ε, τις ψηφοφορίες σας, αλλά 7 λεπτά θα μείνω μαζί σας. Ξέρω ότι έχετε σημαντικά πράγματα να ψηφίσετε. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν μπορούσα να συναντήσω τα μέλη της αντιπροσωπείας που θα μας εκπροσωπήσουν ε, στην συνδιάσκεψη για το κλίμα στο Κανκούν ε, την προηγούμενη Τρίτη. Ήταν όμως, είχαμε το θέμα του προϋπολογισμού και είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ήμουν και ε, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας για, τις, για τη συνδιαλλαγή και ήταν πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα που, με τα οποία έπρεπε να συνδιαλλαγούμε με το Συμβούλιο. Από την άλλη πλευρά προείδρευσα την ε, τελευταία συνεδρίαση στο Στρασβούργο, ε, δεν μπόρεσα να προεδρεύσω ε, για το στο Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, για τα θέματα του περιβάλλοντος, γιατί ακριβώς υπήρχε η διάσκεψη των Προέδρων που ασχολήθηκαν με τα θέματα προϋπολογισμού η, η Επίτροπος, η κυρία Χάντεγκέρδα, που είναι υπεύθυνη για τα θέματα περιβάλλοντος, ε, συναντήθηκε μαζί μου και συζητήσαμε τα πιο σημαντικά θέματα, τα οποία τα γνωρίζετε εξίσου καλά όσο και εγώ. Και το πιο σημαντικό θέμα, το οποίο βρίσκεται επιτάπητος αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την άποψή της Επιτρόπου, είναι η τα μέτρα προσαρμογής των κλιματικών αλλαγών, τα θέματα δασών, ε, τεχνολογία, μεταφορά τεχνολογίας και θα ήθελα να ε, τονίσω ότι όχι μόνο από τις αναπτυσσμένες προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και μεταφορά τεχνολογίας ανάμεσα στις όμενε χώρε ε, και τι αναπτυγμένε χώρε ανάμεσα στι αναπτυγμένες χώρε, Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μεταφερθεί η τεχνολογία με την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ, με την Βραζιλία ενδεχόμενα, με κάποιες χώρε που είναι πιο αναπτυγμένε, πιο προηγμένες από κάποιε άλλε. Επίση, συζητήσαμε για τις ε, συμφωνίες μετά το Κιώτο, τις δεσμευτικές συμφωνίες. Ε, το συζητήσαμε με την κυρία Κόνι Χάντεγκαρτ το θέμα του Γιωχάνεσμπουργκ και της ε, κλιματικής διάσκεψης του Γιωχάνεσμπουργκ και όχι τόσο το Κανκούν, διότι πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα μέχρι ότου καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπέγραψα και έστειλα μία επιστολή στον πρόεδρο κύριο Μπαρόζο για τα συμπληρωματικά 17 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι έτοιμα να πάνε στο Κανκούν πέραν της επίσημης ε, ε, αντιπροσωπείας που είναι 15 ε, μέλη, έχουμε άλλα 17 και θέλουμε και για αυτά τα 17 να υπάρξει διαπίστευση δεν θα είναι μέλη της επίσημης αντιπροσωπείας και το συμφωνήσαμε αυτό εκ των προτέρων. Είναι μια απόφαση των, της διάσκεψης των προέδρων. Στην πλειοψηφία αποφασίσαμε, ε, με πλειοψηφία στη διάσκεψη των προέδρων αποφασίσαμε ότι είναι μεν τα μέλη αυτά θα αποκτήσουν διαπίστευση, όμως δεν θα αποτελούν ε, επίσημα μέλη της ε, αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην επίσημη αντιπροσωπεία όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συμμετέχουν τα 15 μέλη, τα αρχικά, που θα μας εκπροσωπούν στις ε, συναντήσεις με τον τύπο κτλ. Θα εκπροσωπούν την άποψη του Ευρωπα... της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σας πω ότι διάβασα το τελευταίο μας ψήφισμα στο σημείο 79, είναι δικό μου, λέει δίνει εντολές στο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαβιβάσει το θέμα αυτό, το ψήφισμα αυτό, ε, στο Συμβούλιο, στι κυβερνήσει κτλ. Και το ψήφισμα αυτό είναι πάρα πολύ καλό, φίλο να ομολογήσω. Τα πάντα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή για το κείμενο αυτό, για αυτή την Επιτροπή, και θα ήθελα επίση ε, να σα ενημερώσω γιατί τι θα κάνω την άλλη εβδομάδα. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα υπάρξει τρίλογο την Δευτέρα και την Τρίτη Δευτέρα και τρίτη, τρίτη της επόμενης εβδομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα είσαι στο Κανκούν βέβαια. Όλοι σα. Τέλος πάντων, 15 συν 17 εννοώ. Θα υπάρξει όμως ένα τρίλογος, ε, Δευτέρα, Τρίτη, η Κορεπέρ είναι την Τετάρτη, η απόφαση για τη Κορεπέρ θα υιοθετηθεί ή όχι βέβαια από την ε, διάσκεψη των Προέδρων την Πέμπτη, άρα την Πέμπτη είναι πολύ σημαντική η διάσκεψη των Προέδρων και η απόφαση του Συμβουλίου θα ληφθεί την Παρασκευή και μετά τα πάντα θα γίνουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Θα μπορούμε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, του Ευρωπαϊκού, της, ε, να το ψηφίσουμε στις 15 του μηνός, στην τελευταία ε, σύνοδο του Στρασβούργου. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Όλος μου ο ελεύθερος χρόνος εκεί αφιερώνεται και φεύγω για να συναντηθώ με τον Πρωθυπουργό Ρούτερ, γιατί πρέπει να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη για να τους εξηγήσουμε τις απόψεις μας, γιατί ε, μοιραζόμαστε αυτή την ευθύνη. Ε, δεν θέλω να κατηγορήσω καμιά χώρα βέβαια, που δεν ήθελε να συμφωνήσει ε, προηγούμενα, διότι είναι και αυτό δυνατότητα που έχουν, γιατί το συμφωνήσαμε. Γι' αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Την επόμενη εβδομάδα θα ήθελα να πάω στο Ηνωμένο Βασίλειο για να έχω και εκεί τις ίδιες συζητήσεις. Επομένω, προετοιμάζω στι αρχέ εβδομάδα τη συνάντησή μου, το ταξίδι μου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη εγώ, αλλά σε εσά εύχομαι κάθε επιτυχία στα σημεία τα οποία είναι τόσο σημαντικά. Δεν θα είναι μια δεσμευτική συμφωνία βέβαια, το οποίο είναι το πιο σημαντικό για μας, όμως θα ληφθούν σημαντικά βήματα για να φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτή την δεσμευτική απόφαση. Καλή επιτυχία σε όλους σας συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Exactly Ακριβώς 7 λεπτά, όπως μας υποσχεθήκατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπούζεκ ε, γιατί ήρθατε εδώ να μιλήσετε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Όλοι διαισθάνονται την ε, ε, δέσμευση που έχει αναλάβει για το κλίμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήρθατε εδώ να μιλήσετε στην Επιτροπή. Έχετε και καλά νέα βέβαια ότι εκτός από τα 15 μέλη της επίσημης αντιπροσωπείας ε, και τα 17 μέλη τα οποία έδειξαν τόσο ενδιαφέρον να πάνε στο Κανκούν θα πάρουν τη διαπίστευση. Τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε κάποιες συζητήσεις ε, κάπως έντονες. Βέβαια ο προϋπολογισμός είναι το κύριο θέμα της Συνόδου του Δεκεμβρίου. Ε, ξέρω ότι πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια, έχετε αναλάβει υποχρεώσεις ε, για να ολοκληρώσετε την ε, υιοθέτηση του προϋπολογισμού. Ε, το Κοινοβούλιο πρέπει να διαβουλευτεί με το Συμβούλιο. 27 κράτη-μέλη, δύσκολο πράγμα. Η ζωή στο Κοινοβούλιο μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά και στο Συμβούλιο πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, σας ευχόμαστε και σε εσά κάθε επιτυχία και πρόεδρο. Είδαμε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε προσεγγίζουν η μία την άλλη. Θα μπορούσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει την πρωτοβουλία και να οργανώσουμε και την ε, διάσκεψη για το κλίμα του χρόνου στο Ιωάννεσμπουργκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ευχόμαστε και σε εσά καλή επιτυχία. Η Οι πρόεδροι είναι πολύ απασχολημένοι. Αυτό όμως μας δίνει και εμάς ένα περιθώριο χρονικό για την ψηφοφορία που θα συνεχίσουμε τώρα. Και είχαμε φτάσει στην τροπολογία 14, συμβιβαστική τροπολογία, την παράγραφο 7, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 132 Παόλο Μπαρτολότσι ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 15 για την παράγραφο 8 ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 145. Νέσο Τσίλβες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 156 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 158 υπέρ.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 Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 183 με προφορική τροπολογία και κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, με την προφορική τροπολογία, όχι καταπίπτει. 184 κατά αποχές εγκρίνεται 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά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 Μετά περνάμε στη συμβιβαστική τροπολογία 2, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται επίσης. Μετά έχουμε τη 19 της Ελένα Αντωνέσκου, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3, ψήφι υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε για την 27. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 28 είναι κάποια γλωσσική αλλαγή, αλλά πρέπει να το ψηφίσουμε. Λοιπόν, 28 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 και 33 μαζί ψήφι υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Καταπίπτει. 32 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34. Κατά τμήματα και προφορική τροπολογία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγκεντρωτική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5. Να ελέγξουμε την ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα τη 47. Ελέγχουμε λοιπόν. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 ψηφί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58, μόνο το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος της 58, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Και οι φιλελεύθεροι στο τέλος της ψηφοφορίας θέλουν να δηλώσουν τη θέση τους για όλες αυτές τις ψηφοφορίες, οι οποίες είναι κατά, φαντάζομαι. 59. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα μόνο, ψήφι υπέρ, για το πρώτο τμήμα της 59. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενδιαφέρον. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68. Φιλίπ Ζουβά υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά. Να το ελέγξουμε. Για την 72 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 30... Εγκρίνεται και περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. 48 υπέρ, μία αποχή, καμία ψήφο κατά. Συγχαρητήρια στην Μαρίζα Ματίας για την έκθεση αυτή. So, für den Präsidenten hatten wir eine halbe Stunde einkalkuliert, äh, der musste Είχαμε υπολογίσει με μισή ώρα για τον πρόεδρο, τώρα μας έχουν μείνει 20 λεπτά. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε στις 10.30 ακριβώς με την ακρόαση της Κατρίνης Ζεσλα Λανέλ για την αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων της Πάρμας. Διακόπτουμε λοιπόν για 20 λεπτά.